Άρχεται η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της 7 η Απριλίου 2010. Έχετε παρατηρήσεις από αυτόν, όχι. Θεωρούνται λοιπόν τα πρακτικά εγκεκριμένα.